αποδεκτές. Από την ΚΟΕ έχω πάρει ε, μία ε, πρόταση ε, να συμμετάσχει η κυρία Νίνες στον, στην Επιτροπή Πολιτισμού. Έτσι λοιπόν η πρόταση αυτή γίνεται επίσης αποδεκτή. Επόμενο σημείο της μερίσιας διάταξης είναι η κοινή